όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σύντομα θα καταθέσουμε προτάσεις για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Τελειώσαμε με αυτή τη συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. Τώρα, έκθεση ματέρα για την κατάσταση των μόνων μητέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας κυρίως τους χειώδεις εισηγητές και όλους τους συναδέλφους που συνέφεραν στον εμπλουτισμό της έκθεσης με νέες ιδέες για να ενισχύσουμε αυτήν την αδύναμη κατηγορία δυνατών που χωρίς να έχουν κάνει την επιλογή είναι μόνες τους στο μεγάλωμα των παιδιών και παράλληλα προσπαθούν να εργαστούν. Αυτές οι γυναίκες που κινδυνεύουν από τη φτώχεια χρειάζονται ενίσχυση από την Ευρώπη. Ε, μεγάλη μου τίμη που ανέλαβα εγώ την ευθύνη για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης σχετικά με τις μόνες μητέρες στην Ευρώπη. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διαπιστώσουμε μέτρα για την ενίσχυση των μονογονικών οικογενειών. Έγινε πριν από μερικούς μήνες μια ακρόαση στο Κοινοβούλιο για να ακούσουμε εμπειρογνώμονες ενώσεων οι οποίοι εργάζονται με τα προβλήματα των μονογονικών οικογενειών, κυρίως των μόνων μητέρων. Συνάντησα ενώσεις που υποστήριξαν αυτές τις μόνες μητέρες στα κρατημέλη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στο Βέλγιο και στο Βέλγιο μπόρεσα να επισκεφτώ προσωπικά μία ένωση όπου βιώνουν, κατοικούν μόνες μητέρες και εκεί είχα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πληροφορίες με την υπεύθυνη αυτής της, ε, αυτού, αυτής της Ένωσης και μπόρεσα να καταλάβω καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτές τις γυναίκες. Και επίσης κατά το ταξίδι μου στη Βαρσοβία με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Γυναικών μπόρεσα να δω πώς ζουν οι μόνες μητέρες στην Πολωνία. Πρόκειται για μια δημογραφική κατηγορία η οποία αγνοείται και είναι διαφορετική η αντίληψη στην Ευρώπη για τις μόνες μητέρες. Στη Νότιο Μεσόγειο όπως Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα γίνεται δεκτό η διευρυμένη οικογένεια να βοηθάει στην, στο μεγάλωμα των παιδιών, των μόνων μητέρων, αλλά στις βόρειες χώρες τα συστήματα welfare της κυβέρνησης βοηθούν τις single μητέρες με πολιτικές κοινωνικής βοήθειας. Στα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης έχουμε ένα mixed πολιτικών έχουμε ορισμένες οι οποίες συνδέονται με το κομμουνιστικό παρελθόν και άλλες οι οποίες έχουν ιδέες, ε, ένα μείγμα μεταξύ βόρειος, Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι μόνες μητέρες όπως ε, στην Εστονία και στη Λετωνία που φτάνει το 9%. Οι σύγκολ μητέρες στιγματίζονται όπως νέες ανεύθυνες ενώ το 85% είναι μεταξύ των 25 και των 64 ετών. Και πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις της ε, κρίσης ε, και επί αυτών των γυναικών, οι οποίες ε, ήδη επιβαρύνονται από τη διαφορά μισθών που οφείλονται στο φύλλο και αυτές οι μητέρες δεν έχουν τη δυνατότητα να φροντίσουν τα παιδιά τους ή να πάρουν δάνεια η υγεία των μόνων μητέρων είναι χειρότερη από ότι των γυναικών με σύζυγο. Έχουν περισσότερο στρες διότι ασκούν ε, αρμοδιότητες δύο γονέων. Δεν έχουν χρόνο για να ξεκουραστούν. Δεν είναι τόσο μορφωμένες όσο οι παντρεμένες και έχουν δυσκολίες πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας. Λοιπόν, τέλειωσα το χρόνο μου, διότι είχα παρουσιάσει μία έκθεση πιο... Α, πρέπει να διακόψω, ωραία πρόεδρε. Η έκθεση είναι γεμάτη νέες πρωτοβουλίες ε, και κυρίως νέους στόχους που θα πρέπει να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι θα πρέπει αυτή η θεματολογία να αποτελέσει προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι ο αριθμός αυτών των γυναικών αυξάνει το λένε και περισσότερο στην Ευρώπη. Ε, ευχαριστώ κυρία Ματέρα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω την κυρία Ματέρα και να την συγχαρώ. Να την συγχαρώ επειδή ε, διεξοδικά σε βάθος ανέλησε όλα αυτά τα προβλήματα. Η κατάσταση των ε, γυναικών που μεγαλώνουν παιδιά μόνες τους ε, συνδέεται και με την φτώχεια, την παιδική φτώχεια κάθε τρίτο παιδί ζει σε καθεστώς φτώχειας ή στην κατάσταση να, εντα, να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία των φτωχών παιδιών και οι μόνες μητέρες όσον αφορά και τις ε, του όρους εργασίας και την σύγκληση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όλα αυτά οδηγούν σε, μια υπαρξιακή, σε ένα υπαρξιακό θέμα επιβίωσης αυτές τις γυναίκες. Αν δεν μπορούν να πετύχουν αυτά, τότε οι στόχοι της ίδιας της πολιτικής απασχόλησης δεν, μπορούν, δεν μπορεί να, οι στόχοι να ευδοκιμήσουν. Και βλέπουμε την φτώχεια που πλήττει αυτά τα παιδιά που εγκαταλείπονται σε ένα καθεστώς φτώχεια Κάτι πρέπει να κάνουμε και με αποφασιστικό τρόπο λοιπόν. Η κυρία Ζαμπόρσκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Επίτροπε. Οι μόνες μητέρες έχουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για τα παιδιά τους. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος που εγκυμονεί να πέσουν σε, στο καθεστώς της φτώχειας, της παινίας. Γι' αυτό υποστηρίζουμε τις προσπάθειες να τύχουν συνδρομής, να τύχουν αρρωγής οι γυναίκες μετά το διαζύγιο ή όταν μένουν, είναι μόνες τους. Είναι και δαπανηρές οι διεργασίες αυτές. Πρέπει κάτι να κάνουμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες γενικότερα, διότι πολλά διαζύγια σημειώνονται λόγω οικονομικών προβλημάτων και προβλημάτων οικονομικών που πλήττουν τις οικογένειες. Πρώτο πρέπει να είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κατανοήσει ότι οι οικογένειες δεν είναι μια ομάδα απλώς ανθρώπων που συμβιώνουν. Ο γάμος δεν είναι κάτι που βρίσκεται στα χαρτιά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να κατανοήσουν ότι δεν είναι θέμα συγκυρίας, δεν είναι σύμπτωση. Όταν ακούμε σήμερα για παράδειγμα διαρκώς ε, τα θέματα ισότητας ε, των φίλων. αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο των μόνων μητέρων και όχι των μόνων πατέρων. Και αυτό κάτι δείχνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ροήτοβα. Σας ευχαριστώ και εγώ πρόεδρε. Θέλω να υποστηρίξω τα, τις προτάσεις και την έκθεση της κυρίας Ματέρα για την κατάσταση των μόνων μητέρων. Θα πρέπει τα κράτη να υιοθετήσουν τα σωστά πρότυπα, τις σωστές προτάσεις ώστε οι μόνες μητέρες να βρουν τη δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να εξεύρουν τη σωστή ισορροπία για τις οικογενειακές και ε, επαγγελματικές τους ανάγκες. Όχι μόνο όμως για τις μόνες μητέρες αλλά και για τα ζευγάρια διότι τα ζευγάρια δεν πρέπει να ε, έχουν αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης ε, ε, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Επενδύσεις στην ε, εκπαίδευση και παιδεία είναι οι καλύτερες επενδύσεις λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές και τις δημογραφικές αλλαγές. Πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Πρέπει να υποστηριχθούν μη κερδοφόρες, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη των μόνων μητέρων και την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Κώστα. Ευχαριστώ. Κώστα παρακαλώ. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την ενδιαφέρουσα και πλούσια έκθεσή της. Πάνω από 5% του γυναικείου πληθυσμού στην Ευρώπη είναι single μητέρες και θυμίζω ότι το 85% των μόνων γονέων είναι γυναίκες. Οι μονογονικές οικογένειες πρέπει να καλύπτονται από τις πολιτικές εργασίες, κοινωνικές πολιτικές. Το λέει στην έκθεση, πρόκειται για ε, γυναίκες οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Ας πούμε στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε single μητέρες, στην Σκανδιναβία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ στο Νότο κυρίως οι μόνες μητέρες είναι αυτές οι οποίες ε, είναι μόνες μετά από χειρία, διαζύγιο ή χωρισμό. Δηλαδή στο βορρά η κατάσταση είναι πιο ε, προχωρημένα τα, πιο προχωρημένο το φαινόμενο welfare για την προστασία των μόνων μητέρων διότι και ο οικογενειακός ιστός είναι πιο αδύναμος από ότι στο νότο όπου το welfare είναι μειωμένο γιατί, γιατί υπάρχει αυτός ο οικογενειακός ιστός που προστατεύει. Πρέπει λοιπόν εμείς να συγκρίνουμε τα συστήματα welfare και τις καλύτερε πρακτικές για να δούμε ποιο είναι το καλύτερο μείγμα υπηρεσιών που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε ώστε να προβλέπουμε και μη αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και καλύτερη κατάρτιση για να έχουν την πρόσβαση. Η κυρία Φλασίκοβα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Σε πολλές κοινωνίες ιδιαίτερα όσον αφορά τα πατριαρχικά πρότυπα πατριαρχικής κοινωνίας οι μόνες ε, μητέρες ε, δεν την χάνουν του σεβασμού που θα έπρεπε θεωρούν ότι ζουν σε μια μεταβατική περίοδο μέχρι ότου βρουν έναν ε, συμβίο, παντρευτούν και ζήσουν μια ζωή ως σύζυγοι. Πρέπει όμως να ανταποκριθούμε αλλάζοντας πολιτικές σε σχέση με το πρόβλημα των μόνων μητέρων. Είναι ευθύνη των κρατών να βοηθήσουν τις μόνες μητέρες να δημιουργήσουν μια αυτοτελή ζωή, ανεξάρτητη ζωή για αυτές και τα παιδιά τους. Δεν παίρνουν επαρκείς μισθούς, δίκαιους μισθούς και πρέπει να υπάρξουν πολιτικές, κρατικές πολιτικές όσον αφορά την εκπαίδευση, την παιδεία, την κατάρτιση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, την απασχόληση, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στέγασης που θα συνεπικουρούν αυτές τις γυναίκες ή τις οικογένειες, μόνο γονεϊκές οικογένειες. Ευχαριστώ. Grazie. La parola all'onorevole Nevedalova. Κυρία Νεβεδάλοβα. Ναι. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση των μόνων μητέρων στην Ευρώπη είναι φρικτή. Υπάρχει υψηλότατος αριθμός μόνων μητέρων που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ε, ανεργία, πολύ κακή φυσική κατάσταση. Αυτές οι γυναίκες αντιμετωπίζουν <clears throat> κάθε είδους αρνητική διακριτική μεταχείριση. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα που θα υπάρξουν για να τις υποστηρίξουμε, να τις υποστηρίξουμε αυτές και τα παιδιά τους και στη σταδιοδρομία τους, να υπάρξει συμβουλευτική αρρωγή προς τις γυναίκες αυτές και να προσφέρουμε και δυνατότητες για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μόνες μητέρες στα στελέχη στο προσωπικό τους και ε, εκστρατείες που βοηθούν τις μόνες μητέρες δεν έχουν όμως επαρκή χρηματοδότηση αυτές οι πρωτοβουλίες και εκστρατείες. Πρέπει να δούμε και το θέμα της πρόνοιας ή πρόληψης, δηλαδή να ενημερώνονται οι νέοι εκ προημίου όσον αφορά την σεξουαλική τους συμπεριφορά και είναι κρίμα το ότι δεν συμμετέχουν άντρες σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. La parola Η κυρία Τσέσκοβα. Ε, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σκιώδης εισηγήτρια ήμουν εξ ονόματος ε, της ΙΣΙΑΡ ε, της ομάδας μας, σε σχέση με το θέμα της έκθεσης Υπό την αρμοδιότητά μου αυτή θα ήθελα να πω τα εξή. Στη δημοκρατία της ε, Τσεχίας ένα από κάθε τέσσερα παιδιά ζει σε οικογένεια μονογονεϊκή μονογονικών γονέων, μονογονικές οικογένειες. Η πλειοψηφία είναι μόνες μητέρες. Γι' αυτό υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες πολιτικών που θέλουν να βοηθήσουν να εξευρεθεί σωστή ισορροπία σε σχέση με τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές. Ελαστικό ωράριο απασχόλησης, μερική απασχόληση, η εργασία κατοίκων είναι πολύ σημαντικά θέματα. Η υποδομή επίσης για τη μέρημνα των παιδιών είναι σημαντική υπόθεση, κάτι το οποίο διευκολύνει τις ε, μητέρες μητέρες, τις μόνες μητέρες, τις γυναίκες αυτές να, να εργαστούν. Στα θέματα αυτά έχει κέρια σημασία να καταστεί εφικτό να μπορούν να εργάζονται οι μόνες μητέρες και να φροντίζουν τα παιδιά τους όπως ε, πρέπει. Ευχαριστούμε για αυτή την έκθεση. Το έργο της εισηγήτριας ε, είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ε, φυστά την προσοχή στα κυριότερα προβλήματα και καθιστά σαφή στους πιο σημαντικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Είμαι μέλος όμως από την άλλη πλευρά της ε, ECR της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και έχω και μία ερώτηση που θα ήθελα να διατυπώσω. Σε σχέση με τα μέσα, τα εργαλεία που διατυπώνονται στην έκθεση στον τομέα των υγειονομικών, της προστασίας της υγείας και των σχετικών υπηρεσιών, αυτά θα έπρεπε να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεωτικά. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ρυθμίζουν αυτά τα θέματα από πλευράς. Τελευταία τοποθέτηση η κυρία Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε στην Ευρώπη όλο και περισσότερες μόνες μητέρες μεγαλώνουν παιδιά αλλά και μόνοι γονείς πατέρες μεγαλώνουν έτσι τα παιδιά τους χωρίς ιδιαίτερη προστασία Τη οποίας την χάνουν. Όμω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι θα έπρεπε να πει για την κατάσταση αυτών των ανθρώπων που μεγαλώνουν τα παιδιά του αβοήθητοι και αβοήθητες μόνοι και μόνε του. Είναι σημαντικό να βοηθηθούν οι μητέρε και οι πατέρε και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά του. Η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει περισσότερα προγράμματα για την υποστήριξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τη απασχόληση αυτών των ατόμων. Να μάθουν να αποκτήσουν προσόντα και δεξιότητε να μπορέσουν ως ε, ε, ανεξάρτητοι ενδεχόμενα να εργαστούν, ανεξάρτητοι επαγγελματίες, θα πρέπει οι μόνοι πατέρες και μητέρες ε, που μεγαλώνουν παιδιά να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί όσον αφορά την αγορά εργασίας. Ανέφερα τους μόνους πατέρες στην περίπτωση της παρέμβασής μου, διότι πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να αφορά και τους μόνους πατέρες που μεγαλώνουν παιδιά, παρότι ο αριθμός τους είναι πολύ μικρότερος από εκείνος των μόνων, από κοινό των μόνων μητέρων. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος Ρέντινγκ έχει τον λόγο τώρα παρακάτω. To... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Ματέρα. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη και χρήσιμη η συνεισφορά της ε, διότι έχει, σημα... έχει ιδιαίτερη σημασία το θέμα που επέλεξε. Γνωρίζουμε ότι η δομή των νοικοκυριών τροποποιείται συνέχεια στην Ευρώπη και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Εντάξει, υπάρχουν και άντρες, αλλά σε συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται για γυναίκες και είναι αυξανόμενο το ποσοστό τους. Ε, μία πρόσφατη μελέτη του ΩΣΑ δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες σε όλα τα κρατημέλη για αυτό το θέμα. Μέχρι το 2030 προβλέπεται ότι θα σημειωθεί αύξηση ε, από 22-29% των μονογονεϊκών ε, οικογενειών σε σχέση με σήμερα. Οπότε σήμερα βιώνουμε μόνο την ε, αρχή μιας πάρα πολύ σημαντικής τάσης και φυσικά θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Η πρώτη δράση εγγράφεται στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 με στόχο να μειώσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που κατά 20 εκατομμύρια που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικής αποξένωσης. Ε, το αριθμός των παιδιών ε, που ζουν υπό αυτές ε, τις συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει το 30% για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Καταλαβαίνετε ότι μετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ένδυας και κοινωνικού αποκλεισμού και θα θέλαμε μέσα στη στρατηγική του 2020 να προτείνουμε στήριξη προς αυτές τις οικογένειες σε πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ε, δηλαδή περίθαλψη, παιδεία, ε, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τα παιδιά, για τις ε, γυναίκες και για τους άντρες που συντηρούν μονογονιακές οικογένειες και δυσκολεύονται ε, να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας χωρίς να πέσουν στην παγίδα της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και θέλουμε να αποφύγουμε τα λάθη και γι' αυτό συλλέγουμε δεδομένα για να εντοπίσουμε τις ε, τρέχουσες τάσεις εν μέρη στη βάση δεδομένων για τις οικογένειες έτσι ε, όσα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρεπιπτόντως υπάρχουν εν μέρη τα στοιχεία και υπάρχει ένα εργαλείο υπολογισμού τόσο ώστε ε, να συγκρίνουμε τα εισοδήματα διαφόρων οικογενειών. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Οικογένειες είναι μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ε, βέλτιστης, ε, βέλτιστων εμπειριών και εκμάθηση ε, για αυτό το θέμα. Επίσης υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Δύο Φύλων που αναλύει αυτά τα δεδομένα και εκπονεί μεθοδολογία και εργαλεία για την ένταξη του θέματος ε, της ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανταλλαγή των βελτίστων εμπειριών. Ε, Πρόεδρε, είναι πρώτη φορά που σχολιάζουμε αυτό το ζήτημα στην Ολομέλεια και είμαι πεπισμένη ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, έληξε η συζήτηση, θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. Έκθεση της κυρία